Και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη προβλέπεται η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για τη χρήση οπλισμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών. Θα δώσω λοιπόν εκ νέου το λόγο στον Υπουργό Κούρκουλα εξ ονόματος της Αντιπροέδρου Άστον. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, RPA, που είναι ο όρος που συνήθως χρησιμοποιούμε για τα drones, αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, είναι πολύ επίκαιρα και αυτό και λόγω των πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου. Αλλά οποιαδήποτε συζήτηση για επλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα πρέπει να γίνει με βάση με ένα ιστορικό πλαίσιο, γιατί η χρήση τους και οι εφαρμογές τους θα αυξηθούν. Έχουν περισσότερη αντοχή και εν γέννη είναι πιο πολύμορφα στη χρήση τους από ότι τα συμβατικά αεροσκάφη, ε, τα επανδρομένα αεροσκάφη, πράγμα το οποίο θα καταστήσει τη μελλοντική τους χρήση σε μεγαλύτερη κλίμακα αναπόφευκτη. Η συζήτηση για την αυξανόμενη ποικιλία των δυνητικών χρηστών έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και καιρό και έχει γίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη. Τα RPA δεν παίζουν μόνο επιθετικό ρόλο, με το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων τους μπορούν να συμβάλλουν σε διάφορες επιτυχίες στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων. Στο στρατιωτικό τομέα ορισμένα τέτοια αεροσκάφη είναι σχεδιασμένα ώστε να κάνουν ε, κρούσεις, όμως ευρύτερα χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν το σχεδιασμό, την διεξαγωγή και την αξιολόγηση επιχειρήσεων μέσω των αναγνωριστικών τους ε, και δικών του δυνατοτήτων. Καλύτερη εποπτεία σημαίνει τον εντοπισμό απειλών εγκαίρω, ε, αλλά και ε, ενδεχομένω την ε, εξοικονόμηση ζωών των ε, στρατιωτικών. Ε, η εποπτεία σημαίνει εποπτεία για πυρκαγιές, για έλεγχο ε, του βαθμού της πιστοποίησης και ούτω καθεξής. Επιπλέον, οι ιδιωτικές εταιρείες εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης των μη επανδρομένων αεροσκαφών ως τμήμα της, των υπηρεσιών διανομής τους. Θα αυξηθεί λοιπόν η ποικιλία των χρηστών και μιλάμε για τεχνολογίες που εξελίσσονται ταχύτερα ταχύτατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος οικονομικός ε, παράγοντας και εσωτερική αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων ε, με μεγάλο μερίδιο του ΑΕΠ παγκοσμίω θα πρέπει να παίξει έναν ρόλο η ίδια σε σχέση με αυτό το νέο προϊόν και τη νέα τεχνολογία. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όλο ένα και περισσότερο ε, βλέπει να τη ζητάτε να παίξει ηγετικό ρόλο στις ε, επιχειρήσεις επίλυσης κρίσεων και σε αυτές που περιλαμβάνουν στρατιωτικό σκέλος. Ας πούμε η επιχείρηση Αταλάντη είναι ένα σχετικό παράδειγμα. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με τη μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι σαφή ότι θα πρέπει δηλαδή να αυξηθούν οι δυνατότητες των μη επανδρομένων αεροσκαφών, για ε, αποστολές ε, ΚΕΠΑ για, για τη βελτίωση της ε, ε, της, ε, της στρατηγικής περί ναυσιπλοείας. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τέτοια προϊόντα, να αποφασίσουμε μάλλον ε, πολιτικά αν θα χρησιμοποιήσουμε ξένη τεχνολογία ή θα επιλέξουμε τη δική μας τεχνολογία. Αυτή θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της Ένωσης για θέματα ασφαλείας αλλά και θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Τα θέματα που σχετίζονται με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ε, εμπίπτουν σε διάφορε αρμοδιότητε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη 19η Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου ήταν ευκαιρία για καποια καθημερινά να εξετάσουν τι είδου δυνατότητε μη επανδρομένων αεροσκαφών μπορεί να χρειαστούν υπό την αιγίδα τη ε, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αμήνης μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο 2020-2025. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε εντολή επίση για εναρμόνιση ανάμεσα στους θετικού και πολιτικούς χρήστες όσον αφορά την ένταξή του στην αέρια κυκλοφορία αλλά και την αντοχή τους και το βεληνικές τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ασφάλεια αλλά και ε, ε, βεληνικές όσον αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που θα χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο μας. Επίση, υπάρχουν κάποιε ανησυχίε όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνού δικαίου. Η χρήση των μη επανδρομένων σκαφών, αν και η ε, αναχέτηση τη τρομοκρατία έχει ήδη θυγεί από τον ειδικό εισηγητή για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, η θέση μα ωστόσο είναι ξεκάθαρη ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πω οποιαδήποτε χρήση θα είναι συνεπή τόσο με το ευρωπαϊκό όσο και με το διεθνέ δίκαιο δεν πρόκειται για την τεχνολογία αλλά για τη χρήση αυτής που είναι το θέμα κλειδί. Εδώ συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα. Εν τω μεταξύ, η ΕΠΑ είναι η ε, πρωτοπόρος στην παραγωγή και χρήση των RPA, ενώ πολλές άλλες χώρες όπως η Ισραήλ, η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν, ο Ισημερινός αναπτύσσουν δικό, δικές τους εθνικές δυνατότητες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου έδωσε επίση εντολή για τη διερεύνηση μια τέτοια αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Ξεκινάμε τη διερεύνηση του πώ θα ικανοποιήσουμε τι προτεραιότητε τη Ένωση, πώ θα παίξουμε τον ρόλο που μα αντιστοιχεί στον κόσμο, θα ικανοποιήσουμε τι αγορέ μα, τι δικέ μα απαιτήσει, αλλά και πώ θα ενισχύσουμε τη βιομηχανική μας βάση. Η πολιτική μας απόκριση σε όλες αυτές τις διάφορες πτυχές της κρίσης RPA θα εξελιχθεί όταν θα γνωρίζουμε καλύτερα ότι αυτοί που θα οδηγήσουν όλες αυτές οι εργασίες και αυτή η τεχνολογία. Γνωρίζουμε πως ε, θα υπάρξουν προκλήσεις στο μέλλον και ότι πρέπει να εξετάσουμε διάφορες πτυχές. Γι' αυτό και προσβλέπω στην απόψινή συζήτηση και ε, να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ. Grazie. Ε. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχουν οι ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Εξ του ΕΛΚ, ο κύριος Γκάλερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε από το Συμβουλίο για τη δήλωσή σας με την οποία και συμφωνώ πλήρως. Είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων για αυτό το οποίο είπατε ευθύ εξ αρχή, πω η τεχνολογία των μη επανδρομένων αεροσκαφών έχει ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών και στον πολιτικό τομέα, κυρίω στον πολιτικό τομέα, αλλά και στον στρατιωτικό. Εμείς ως ομάδα του ΕΛΚ θα θέλαμε ένα ψήφισμα το οποίο θα αντικατόπτριζε ακριβώ το εύρος αυτού του φάσματο. Δεν καταφέραμε να το περάσουμε παρόλα αυτά. Όμως σε ένα πνεύμα συμβιβασμού θα έλεγα καταλήξαμε σε αυτό το κοινό ψήφισμα. Όπως ήδη έχω πει για την ευρωπαϊκή βιομηχανική και αμυντική βάση θεωρώ πως ε, χρειάζεται για τις ε, επιχειρήσεις ΚΕΠΑ να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και συγκεκριμένα οι δυνατότητες ε, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ο δε στρατηγός Ντέρος ο επικεφαλής ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Επιτελείου στην Επιτροπή την Υποεπιτροπή με ασφάλειας και άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε πως θα έπρεπε να στηριχθούμε και σε αυτά τα μέσα. Επίσης και τα οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων των στρατιωτών μας. Δεν βλέπω δε όσον αφορά το νομικό πλαίσιο καμία πιθανότητα παράνομης χρήσης τους. Επίσης ξεκαθαρίζουμε βεβαίως με αυτό το ψήφισμα πως είμαστε κατά των πλήρως αυτοματοποιημένων τέτοιων αεροσκαφών και πράγματι πρέπει να τα χειρίζονται άνθρωποι και να μην ε, επαφίεται η λειτουργία τους μόνο σε έναν αλγόριθμο. Οπότε συμφωνούμε και σε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τους σοσιαλιστές, ε, η κυρία Γκόμες για μισή λεπτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο τα μη επανδρομένα οχήματα ε, χρησιμοποιούνται από μεγάλες δυνάμεις όπως η ΕΠΑ. Ε, πέρα από το νομικό πλαίσιο και μέσα στα πλαίσια εμπολέμων καταστάσεων. Για μια τέτοια τεχνολογία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να έχουμε εγγυήσεις για την σωστή χρησιμοποίησή τους. Όταν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι παράνομη η χρήση τους και δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό τη στιγμή που τα κράτη-μέλη θα ε, ενισχύσουν αυτή την τεχνολογία θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για την χρήση των ε, drones και να είμαστε υπεύθυνοι μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και του διεθνές ε, ποινικού δικαίου. Μέσα στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το δικαίωμα στη ζωή αποκλείοντας την χρήση των drones πέρα από τις εμπόλυμες καταστάσει. καταστάσεις και δεν θα πρέπει να υπάρχει εξωεδαφική χρήση τους γιατί θεωρείται εγκληματική πράξη και είναι κολάσιμη γι' αυτό το λόγο. Επειδή είναι μία τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται από μακριά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει την τεχνολογία αυτή στις διεθνείς συμβάσεις τι θα κάνουμε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιήσουν έξω ή ενδοεδαφικά. Ευχαριστούμε πολύ από τους φιλελεύθερους, κυρία Λάτφορντ, για δύο λεπτά. Ε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλέ στοιχεία που μα ανησυχούν όσον αφορά τη χρήση αυτών των δρασκόμενων για να σκοτώνει τον κόσμο. Γιατί ε, πρόκειται για μη παντρωμένα και οπλισμένα. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά το, τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και όπως προανέφερε η κυρία Γκόμες απαγορεύονται για ε, ανθρωποκτονίες εκτός δικαστικών αποφάσεων. Χωρίς το σπάνιο προηγουμένη διχαστική απόφαση και οπότε δεν θα πρέπει ακόμα και σε ε, πολέμους να είναι στόχοι οι άμαχοι. Πριν από ένα χρόνο είχαμε πει ότι πρέπει να περιορίσουμε τις περιπτώσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα αεροσκάφη εκτός των εμπορικών ζωνών, αλλά τέλο πάντων ούτε αυτό για την υποθεί και τη σαφήνεια και αυτό είναι ένα μέρο τη όλης προβληματική για το ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα, δεν υπάρχει διαφάνεια και η CIA δεν επιβεβαιώνει, τέλο πάντων αρνείται ότι τρέχει ένα τέτοιο πρόγραμμα για τέτοια αεροσκάφη, αλλά ε, όπως η πει και οι και οι υποφαινομένοι, ότι σε κάποια μυστική υπηρεσία να θέτουμε μια τέτοια εκστρατεία ενώ χρειάζεται διαφάνεια θα πρέπει να υπάρχει ένα κατόφλεπο. Ένας όσον αφορά ε, το, το ότι θα πρέπει αυτά να είναι μόνο η τελευταία λύση εδώ τέλος αεροσκάφη επίσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από ποιον να είναι γιατί έτσι και η Αλκάιντα θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει πέραν από τι δυτικέ κυβερνήσει. Και κάποιοι τρομοκράτε που το κάνουν αυτό, θα πρέπει να τραβήξουν την κόκκινη γραμμή τώρα. Χρειαζόμαστε μια ενωσιακή πολιτική ε, για τέτοιου είδου ε, επιδρομέ αυτών των αεροσκαφών και θα πρέπει επομένω να αποφύγουμε ένα νέο σκάνδαλο ε, παρανομία, ε, και η ε, ευρωπαϊκή συνενοχή ε, αυτό μας κάνει συνένοχος, οπότε δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Από τους Πράσινους, η κυρία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Προεδρία του Συμβουλίου και την Κομισιόν για την δήλωση. Έχει φτάσει η στιγμή να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ιδρύθηκε προσφάτως ε, μια ομάδα 7 κρατών μελών με στόχο να αναπτύξουν τέτοια αεροσκάφη κάτι το οποίο χαιρέτησε και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία. Θα πρέπει βεβαίως να δούμε με την πρακτική των ΙΠΑ. Επί Προέδρου Ομπάμα ανέβηκε κατακόρυφα ο αριθμός των επιθέσεων με τέτοια αεροσκάφη. Υπάρχουν λοιπόν ηθικά ζητήματα και νομικά ζητήματα, καθώς γίνεται η, ε, το να σκοτώσει κάποιον τόσο εύκολο ώστε δεν το σκέφτονται πλέον χώρες όπως το Πακιστάν, η Εμένη ή η Σομαλία δεν είναι επισήμως θέατρα επιχειρήσεων πολεμικών και εκτός ε, θεάτρων πολεμικών επιχειρήσεων απαγορεύεται να σκοτώνει κανείς. Πρόκειται για έναν γενικό λόγο πόλεμο κατά τη τρομοκρατία και η χρήση του αποτελεί τμήμα αυτού του πολέμου. Εγώ το θεωρώ λάθο. Αλλά και αν υποθέσουμε πω ισχύει κάτι τέτοιο, ακόμη και τότε ε, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Στο δικό μα το ψήφισμα μιλάμε για το νομικό πλαίσιο για την χρήση οπλισμένων τέτοιων αεροσκαφών. Εμεί ζητάμε να μην χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για εξοδικαστικέ και και εξοεδαφικές επιχειρήσεις. Η χρήση τους λοιπόν θα πρέπει και η παραγωγή και εξαγωγή τους θα πρέπει να υπόκειται σε ε, όλες τις σχετικές διατάξεις ε, και για την εξαγωγή όπλων και να οδηγηθούμε σε μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση τους. Και είναι αυτονόητο βεβαίως πως ζητάμε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πλήρως αυτόματα συστήματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση τα οποία θα λαμβάνουν την απόφαση να σκοτώνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, Σας ευχαριστώ, Λούζινγκ, για την ΚΟΕ για δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω πως η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου συμφωνεί πως η στοχευμένες εξοδικαστικές εκτελέσεις πρέπει να απαγορευτούν. Το ότι οι οπλισμένοι, τα οπλισμένα μη πανδρομένα αεροσκάφη πρέπει να υπαχθούν στο καθεστώς εξοπλισμών και εξαγωγών οπλικών συστημάτων. Αυτό είναι βεβαίως θετικό γιατί πέραν από την ε, ηθική διάσταση δεν υπάρχει καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Βεβαίως εδώ πέρα από το Κοινοβούλιο δεν είχαμε μια καταδίκη επί τη αρχής της χρήσης τους. Οι επιθέσει αυτέ δεν εμποδίζουν ούτε τι τρομοκρατικέ επιθέσει, ούτε τους, τρομοκράτε, Σκοτώνουν. Σκοτώνουν αμάχους οι οποίοι μάλιστα δεν κατονομάζονται ω τέτοιοι αλλά λέγονται παράπλευρε απώλειες. Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν μπορεί κανεί σε αυτές τις χώρε να πάει ούτε σε γάμο, ούτε σε κηδεία, ούτε στην αγορά. Δεν δικαιολογείται αυτό με τίποτα. Δεν καταπολεμάται η τρομοκρατία με τρομοκρατία. Τα, οι στόχοι του διεθνούς δικαίου μπορεί να επιτευχθούν μόνο με τα ανάλογα μέσα. Εδώ πέρα δολοφονούνται πολίτες, υπονομεύεται η δημοκρατία και ρίχνουν πάρα πολύ χαμηλά το κατόφλι της βίαιης επέμβασης αλλά βεβαίω πρόκειται για έναν βομβαρδισμό, μια τεχνολογία βομβαρδισμού, η οποία βεβαίω χρηματοδοτείται εδώ πέρα με κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί ζητάμε την απαγόρευση των πολεμικών μη επαναρμένων αεροσκαφών, ακόμα και αν δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Σήμερα ελπίζω να είναι δυνατόν στο προσχέ μέλλον από την ομάδα της Ελευθερίας και Δημοκρατίας ο κύριος Τέρο για ένα λεπτό. Ένα λεπτό με συγχωρείτε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η χρήση των ε, drones αυτή η νέα τεχνο... πρόκειται για μια νέα τεχνολογία, κάτι το ναι. οποίο δεν αμφισβητείται και χρησιμοποιείται από ε, διάφορες ε, από διάφορες ένοπλες δυνάμεις και σε εμπόλεμες καταστάσεις. Όμως δεν νομίζω ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι νέα και δεν ε, βλέπουμε, δεν μπορούμε να δούμε κατά πόσο δεοντολογικά κάτι τέτοιο αιτιολογείται. Είτε πρόκειται για ε, ε, επανδρομένα είτε για μη επανδρομένα. Οι παράνομες δραστηριότητες είναι παράνομες. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς προωθείται η χρήση των όπλων. Όμως δεν αλλάζει η φύση αυτών των δράσεων. Στάντλερ, για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα γιατί πρέπει να γίνει. Γιατί οι δυνατότητες που έχουν μυστικές υπηρεσίες για τη χρήση τέτοιων μέσων αυξάνονται. Βλέπουμε πως χρησιμοποιούνται ε, ελεύθεροι σκοπευτές στη Βενεζουέλα, στη Δαμασκό, στο Κίεβο. Έτσι ανάλογα έχουν κάποιες υπηρεσίες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μη επανδρομένα αεροσκάφη και αυξάνεται ο αριθμός των αμάχων θυμάτων. Και κοινικά τους λέμε παράπλευρες απώλειες. Αυτός ο κινησμός πραγματικά δεν συμβιβάζεται με τις αξίες τι οποίε λέμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε. Αυτό ισχύει για αυτή την περίπτωση. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται αυτά τα αεροσκάφη για να εκτελέσουν θανατικές ποινές που δεν έχει εκδώσει κανένα δικαστήριο παρά μόνο μυστικές υπηρεσίες. Γνωρίζουν δε οι χειριστές τους πως σκοτώνονται αθώοι άμαχοι και γνωρίζοντας πως τελικά πρόκειται μόνο για άσκηση πολιτικής ισχύω. Και αν εδώ πέρα δεν μιλήσει ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε πλέον το ηθικό ανάστημα για να πούμε οτιδήποτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζεκ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Πολωνία λέμε ότι καμιά φορά κανείς κάνει ό,τι πρέπει από το χέρι του. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέρει αυτό το οποίο θέλει. Βλέπουμε ότι αυτά τα αεροσκάφη, τα μη επανδρομένα χρησιμοποιούνται κάθε μέρα. Έχουμε 80 χώρε σε όλο τον κόσμο που τα χρησιμοποιούν. Βεβαίω, τα περισσότερα από αυτά τα κράτη δεν χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, τα μη επανδρομένα για στρατιωτικού σκοπού. Το κάνουν, α πούμε, για να προστατεύσουν τα σύνορα ή το κάνουν για κάποιες κατεπίγουσες περιπτώσεις, ή κάποιες διασώσεις κατά θάλασσα και σε κάποιες άλλες περιστάσεις που θα μπορούσαμε να τις περιγράψουμε ως ε, μη στρατιωτικές ε, επιχειρήσεις. Και έχουμε βέβαια ο, από αυτά τα 80 κράτη περίπου τα 20 τα οποία χρησιμοποιούν για στρατηγικού σκοπού αυτά τα αεροσκάφη. Στην πράξη πάντω κυρίω η χρήση γίνεται από ΙΠΑ και Ισραήλ. Μα ε, δημιουργούνται ανησυχίε και θεωρούμε ότι θα πρέπει ε, να υπάρξει ε, νομοθέτηση, περιχαράκωση του υπό ποιου χρησιμοποιούνται αυτά τα αεροσκάφη, γιατί προς το παρόν δεν συντρέχει κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να προβούμε σε τέτοια ρύθμιση των νωρίτερο δυνατόν. Πάντοτε υπάρχουν παραπλευρές απώλειες όπου χρησιμοποιούνται αυτά τα αεροσκάφη. Γι' αυτό δεν είναι αποδεκτό. Πάντω, αν δείτε τι γίνεται με τα συμβατικά όπλα, στου διάφορου ε, πολέμου ε, του 20ου αιώνα και τότε είχαμε παραπλευρές απώλειες. Ευχαριστούμε η κυρία Κοπά για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα βρισκόμαστε πλέον πολύ κοντά σε μια εποχή όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα αποτελούν μέρος της αμυντικής υποδομής κάθε κράτους. είναι λοιπόν αναγκαίο η ευρωπαϊκή ένωση να έχει μια κοινή πολιτική για το πλαίσιο χρήσης τους. επικρατεί άποψη ότι τα αεροσκάφη αυτά αποτελούν εργαλεία ειρήνης και ασφάλειας. αναμφισβήτητα η χρήση τους είναι πολυδιάστατη και εξαιρετικά ωφέλιμη σε πολλούς τομείς εκτός της αμυντικής λειτουργίας όπω για παράδειγμα τη χαρτογράφηση, του συνοριακού ελέγχου τη καταπολέμησης πυρκαγιών και της αγροκαλλιέργειας. Δυστυχώ όμω την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε την ευρεία χρήση ενόπλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εξοδικαστικές στοχευμένε δολοφονίες στα εδάφη τρίτων κρατών. Τέτοιε επιχειρήσει πραγματοποιούνται κάτω από ένα πέπλο μυστικότητα, κυρίω από τι Ηνωμένε Πολιτείε και εκτό πλαισίου τη διεθνού νομιμότητα παράλληλα είναι απαράδεκτο έστω και να συζητείται η ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων οπλικών συστημάτων που θα προβαίνουν σε στρατιωτικά χτυπήματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. για να μην επαναληφθούν ανθρωπιστικές τραγωδίες όπως αυτές που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια κυρίως στο πακιστάν και στην ιεμένη η ένωση θα πρέπει φανερά και ξεκάθαρα να αντιταχθεί σε τέτοιες πρακτικές να ζητήσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση των ενόπλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τρίτες χώρες και να καταλήξει μια κοινή θέση σχετικά με τη χρήση τους με γνώμονα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. η στρατιωτική χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών δεν εγείρει νέα πραγματικά ερωτήματα σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο της έναπλης σύγκρουσης. η τεχνολογία δεν είναι το κλειδί για τη λύση του προβλήματος. λύση είναι μόνο η σωστή χρήση της. ευχαριστώ. Ο κύριος Κρόμπεργκ για ένα λεπτό. κυρία, μέχρι τώρα η αγορά των μη επανδρομένων αεροσκαφών δεν ήταν ρυθμισμένη. Πολλά χρήματα έχουν δαπανηθεί και ε, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι πρέπει να δαπανηθούν ακόμα περισσότερα χρήματα. Πριν δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα του φορολογουμένου, για, θα πρέπει να ορίσουμε ένα νομικό πλαίσιο για τη χρήση τους. Χρειαζόμαστε δημοκρατική επίβλεψη και ε, λογοδοσία, καθώς και διαφάνεια και γενικότερα λογοδοσία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το τον ε, αγώνα υπέρ της χρήσης αυτών των όπλων. Θα πρέπει να ενταχθούμε στο διεθνές πλαίσιο ελέγχου της χρήσης όπλων και δεν μπορούμε να δεχτούμε τα όπλα που σκοτώνουν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγκουράκης για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, και μόνο το γεγονός ότι συζητιέται η χρήση των μη επανδρομένων πολεμικών αεροσκαφών αντί να επιδιώκεται η πλήρης απαγόρευσή τους είναι μια ακόμα απόδειξη για τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ένωσης. φαίνεται ότι δεν είναι αρκετοί οι χιλιάδες αθώοι που έχουν δολοφονηθεί ήδη από τα όπλα αυτά μάλιστα και με παράνομες πτήσεις από τις ακτές της σικελίας. η ανάπτυξη νέων δολοφονικών πολεμικών συστημάτων αποτελεί τμήμα των αποφάσεων της συνόδου κορφής της ευρωπαϊκής ένωσης που εντείνουν τον υπεραλιστικό επιθετικότητά της. η ευρωπαϊκή ένωση επιδιώκει να αναπτύξει την κατασκευή και χρήση τέτοιων οπλικών συστημάτων από τι πολεμικέ τη βιομηχανίε και το consortium που προωθούν γαλλία γερμανία ελλάδα ιταλία ολλανδία πολωνία και ισπανία την ανεμπόδιστη χρήση του εναέριου χώρου και την μελλοντική ενεργοποίηση των όπλων αυτών ενάντια και στου λαού των κρατών μελών. δισεκατομμύρια ευρώ από την λαιλασία του λαϊκού εισοδήματο θα κατευθυνθούν στα μονοπόλια τη πολεμική βιομηχανία σε πολεμικά ερευνητικά προγράμματα για την τελειοποίηση των δορυφορικών και άλλων συστημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης που είναι αναγκαία για τα νέα όπλα την ίδια στιγμή που η ευρωπαϊκή ένωση διαλύει την αμυντική βιομηχανία της ελλάδας γιατί δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των μονοπωλίων. τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας όχι μόνο δεν αξιοποιούνται για την ικανοποίηση της λαϊκής ανάγκης αλλά αντίθετα χρησιμοποιούνται στον ανταγωνισμό των υπεραλιστών για κέρδη και επιρροή. Ο κύριος Πρέντα για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είτε μας ενδιαφέρει είτε όχι, τα drones στι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν ε, ένα ε, όπλο το οποίο πραγματικά χρησιμοποιείται. Στην ε, υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάναμε μία επίσκεψη στην Ιεμένη και μεταξύ άλλων μιλήσαμε για τη χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών και είδαμε ότι δεν συμφωνούσαμε όλοι στην υποεπιτροπή για την χρήση αυτών των αεροσκαφών στις ένοπλες δυνάμεις οι πρέσβεις ορισμένων δυτικών χωρών δεν έχουν την ίδια οπτική γωνία. Το λέω γιατί δεν υπάρχει διεθνή συνένεση επί του θέματος. Γνωρίζουμε ότι η μαζική χρήση αυτών των αεροσκαφών εκτός εμπολέμων καταστάσεων μπορεί να βλάψει και να είναι κάτι το ολέθριο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται έξω από ζώνες πολεμικών σειράξεων. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε τους κανόνες χρήσης εκτός εμπολέμων ζώνων, να ορίσουμε νόμιμους στόχους και να υπάρχει διαφάνεια αυτών των επιχειρήσεων μέσα στα πλαίσια της ε, πολιτικής ευθύνης ε, που φέρουμε σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάουιτ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από τρεις μήνες σε αυτήν εδώ την αίθουσα δώσαμε στη Μαράλα Κιουσαφσάη το βραβείο Ζαχάροφ. Ένα θύμα των Ταλιμπάν. Κανείς δεν μπορεί να πει πως είναι υπέρ της τρομοκρατίας ή ο κύριος στρατηγός Μακρίσταλ, πρώην διοικητής των δυνάμεων της ISAF στο Αφγανιστάν. Αυτό που τους ενώνει είναι πως τα χτυπήματα με μια επανδρομένα αεροσκάφη εκτός των ζωνών συγκρούσεων καθιστούν τρομοκρατία πιο πιθανή. Να είμαι σαφής, μπορούν να σώσουν ζωές, εμείς είμαστε υπέρ της ε, έρευνας. Δεν θα μπω εγώ στον αντιαμερικανισμό, αλλά πρέπει να ε, δούμε τις αμερικανικές ε, πρακτικές των λεγόμενων εκτελέσεων και των χτυπημάτων με υπογραφή. Η χώρα μου έχει καταδικάσει τα χτυπήματα αυτά και δεν θέλει να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή ανάπτυξή τους, αλλά με 18 κράτη-μέλη να έχουν τέτοια αεροσκάφη πρέπει το Κοινοβούλιο να τονίσει πως πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και βεβαίω εκφράζουμε την επιφύλαξή μας για πλήρω αυτοματοποιημένα όπλα που δεν χρειάζονται ανθρώπινη παρέμβαση και ζητάμε από τις χώρες εντός και εκτός Ευρώπης να ερευνήσουν τους κανόνες εμπλοκής για την χρήση τους. Ευχαριστώ κύριο Σπάσκου για ένα λεπτό εκτός ε, ε, μικροφώνου. Το 2013 υποστηρίξαμε ε, αυτό το, τα αεροσκάφη μέσα στα πλαίσια του Now it a... από το 20 μέχρι το 25 και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο χρησιμοποιούνται για πολιτικούς ε, σκοπούς. Η αρνητική διαφήμιση σε σχέση με τη χρήση ανθρώπινων στόχων ε, οδηγεί σε μία αντίσταση της χρήσης τους ε, γενικότερα, κάτι το οποίο είναι κατανοητό, γιατί δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι είναι ένας πολύ ε, καλός τρόπος σε περίπτωση ενδυνάμει καταστροφής να, μπορεί να γίνει παρέμβαση για να διασωθούν ζωές ή σε ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις το οποίο όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση και η χρήση αυτών των ε, ε, πανδρομένων αεροσκαφών. Όταν όμως το τζίνι βγει από το μπουκάλι, ε, τότε δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής, ακόμα και αν είναι περιορισμένη χρήση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρλάκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το κοινοβούλιο όμω πρόκειται να τοποθετηθεί κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά αυτό το τα εξοπλισμένα, μη επανδρομένα σκάφη. Και έχουμε αυτό το ψήφισμα, το οποίο θα είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη απαγόρευση τη χρήση αυτών των απαράδεκτων αποθετικών όπλων. Και αν υπάρχει ένα μόνο λόγο για να απαγορεύσουμε για πάντα τη χρήση αυτών των αεροσκαφών, θα μπορούσε να είναι το ότι πρόκειται για ένα νέο όπλο. Εμεί κερδίσαμε το Νόμπελ τη Ειρηνή. Και ένα από του λόγου είναι ότι θέλουμε να ε, φωνάξουμε σταματήστε τα νέα όπλα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία ούτω ώστε να επινοείτε νέα όπλα. Οπότε με εκπλήσουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί που θέτουν ε, τόσοι συνάδελφοι για το ζήτημα αυτό. Το διεθνέ Δίκαιο απαγορεύει τις αφαίρετες ανθρωποκτονίες ε, και αυτό θα πρέπει να είναι επίση, ένα λόγο πέραν των όσων είπαμε πριν θα πρέπει να έχουμε μια ατσάλινη ε, αμεταγίνητη θέση για αυτό το όπλο. Επομένω, πρόκειται τώρα για ένα πρώτο βήμα για την πλήρη απαγόρευση αυτού του όπλου. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch Ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, πρόσωποι του Συμβουλίου, τα μη παντρεμένα αεροσκάφη θεωρούνται ένα δημιούργημα της νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Χρησιμοποιούνται και για στρατιωτικούς και για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούνται επίση σε κάποιε καταστάσει που χροντίζουν κατεπίγουσε όπω πυρκαγιέ ή πλημμύρε. Ε, Ακόμα και οι μετρολόγοι χρησιμοποιούν αυτά τα αεροσκάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινό στρατό. Οπότε δεν μπορεί να απαγορεύσει στα κράτη-μέλη να αποκτήσουν αυτό το όπλο για την άμυνα τους. Θα μπορούσε πάντως να συναυθεί μια ε, συμφωνία, μια σύμβαση ε, διεθνής που να περιορίζει τη χρήση αυτών των όπλων, αυτών των αεροσκαφών, να μην δηλαδή σε περίπτωση πολέμου. Μορβάη. Ευχαριστώ. Βεβαίως υπάρχουν πολύ λίγοι από τους 700 ε, βουλευτές, 700 και κάτι, μιλάμε για πραγματικά ανθρώπινα δράματα και τραγωδίες και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μιλάμε για τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών ως όπλα και αυτό είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα. Ίσως θα πρέπει να διοργανώσουμε και ακροάσεις ή κάποια ακρόαση επί του θέματος γιατί πρόκειται για μια ειδική τεχνολογία. Μπορούμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους στην Ιεμένη που έχασαν τους δικούς τους εκεί βεβαίως γίνεται λόγος για παράπλευρες απώλειες. Θα πρέπει να σταθούμε πολύ περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ε, αεροσκάφη αυτά κατά της τρομοκρατίας, διότι ε, υποθάλπουν την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Grazie. Ε, ora si è concluso il Τελείωσε η διαδικασία Catch the Eye. Το λόγο έχει ο Υπουργό ε, Κούρκουλας ε, εξ ονόματος της Αντιπροέδρου Άστον. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας επί του σημαντικού αυτού θέματος. Εγώ θα τονίσω τα εξής. Πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο θα αναπτυχθεί η πολιτική επί των αεροσκαφών αυτών θα επηρεαστεί από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον από πολιτικούς, πολιτικές παραμέτρους, από τα κράτη-μέλη, θεσμικά όργανα, τους ψηφοφόρους μας, αλλά και από την τεχνολογία και τη βιομηχανία. Βεβαίω τα θεσμικά όργανα μπορούν να καθοδηγήσουν τις αγορές, αλλά θα είναι μια διαδραστική διαδικασία. Οπότε ένα είναι σαφές. Θα υπάρξει μια μεγάλη αγορά για αυτά τα αεροσκάφη. Επίσης, όπως προχωράει, ε, προχωρούν οι εργασίες που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάποια κράτη-μέλη θα σκεφτούν ε, ποια τέτοια αεροσκάφη χρειάζονται, πιθανώς με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσία. Δεν έχουμε φτάσει όμως ακόμα στην φάση λήψη απόφαση για ανάπτυξη τέτοιου αεροσκάφου. Καθώς εξελίσσεται η συζήτηση να θυμόμαστε το πλαίσιο. Πρέπει να δούμε τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο και να αποφασίσουμε το τι χρειαζόμαστε. Θέλω επίση. να αναφερθώ στη μόρφωση με το διεθνέ δίκαιο και να επαναλάβω πως εμείς θεωρούμε πως όλες οι ένοπλες συγκρούσεις πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές και βεβαίως συζητάμε τέτοια ζητήματα με τους διεθνείς εταίρους μας. Επίσης, υπήρξε μια αναφορά στις ηθικές πτυχές της χρήσης τους. Τα ηθικά πλαισία για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν ήδη. Η χάρτα είναι ένα παράδειγμα. Καθώς λοιπόν εξελίσσεται η τεχνολογία, θα εξετάσουμε βεβαίως την συμβατότητά τους με τα μέσα αυτά και ακόμη, και μια φορά, για, ακόμη φορά για την νομιμότητα χρήσης τους. Γιατί τέθη αυτό από πολλούς βουλευτές. Η άποψή μας είναι πως η χρήση τους πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος μετά το πέρας της συζήτησης. Η συζήτηση έχει λήξει και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι.